Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Όσοι δεν έχουν καθίσει, παρακαλώ να καθίσουν για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να καλωσορίσω τους δύο εκπροσώπους της Πολωνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ετούτο το εξάμεινο. Τον κύριο Γέρζι Μίλλερ και τον κύριο Κρίστοφ Κβιατκόφσκι, αν δεν κάνω λάθος την προφορά. Υπουργοί Εσωτερικών και Δημοσίας Διοίκησης και Δικαιοσύνης θα πάρουν το λόγο για να μας παρουσιάσουν την ατζέντα για τους συγκεκριμένους τομείς της Προεδρίας. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μοιραστώ με τους συμμοναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ τα συνήθη. Καταρχάς, έγκρισε τις ημερήσεις διάταξης. Στις 13 Ιουλίου, από τις 12 έως τις 12.30, το σημείο 16 της ενημέρωσης για τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα για τη Συμφωνία Προστασίας των Δεδομένων θα γίνει ε, και κλεισμένο των θυρών. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη και, και προχωρώ στις ε, συνήθεις ανακοινώσεις για τους ε, για τις εκθέσεις και τις νομοδοτήσεις. Ο κύριος Δίας Δεμέρα είναι εισηγητή για την έκθεση ε, των θεωρήσεων για, τις, ε, για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ είναι εισηγήτρια για, το, για την έκθεση για τα ελάχιστα πρότυπα θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Η κυρία Αντωνέσκου είναι εισηγήτρια για την έκθεση του δικαιώματος πρόσβασης σε, δικαι, σε δικηγόρο στις ποινικέ διαδικασίες. Η κυρία Γκυγιόμ είναι η συγγήτρια της έκθεσης για τη διεθνή προστασία. Ο κύριος Μασίπ εγκρίθηκε ως εισηγητής για την έκθεση της, ε, ε, ε για την έκθεση για τους ε, ετούντες ασύλου. Ο κύριος Ρωμέρο Λόπες, ε, εισηγητής για την αμοιβή αναγνώριση προστατευτικών μέτρων σε αστικά θέματα, η κυρία Φλότρ, εισηγήτρια για την έκθεση για την ε, πολιτική γειτονία και η κυρία Σντανόκα, εισηγήτρια για την έκθεση για την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια το 2010. Αντιρρήσεις υπάρχουν? Όχι. Οπότε θεωρούνται εγκεκριμένε αυτές οι εκθέσεις. Πάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Πάμε στο σημείο 4 λοιπόν, κατευθείαν, που είναι το σημείο που αφορά τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα τη δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων. Όπως είπα, είναι μεγάλη μα τιμή και χαρά εδώ να έχουμε σήμερα και τον κύριο Γερζι Μίλλερ, τον ε, Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων και Διοίκησης και τον ε, Υπουργό Κβιατκόφσκι, Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις τους για τους τομείς της ευθύνης τους και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις. Κύριε Μίλλερ, έχετε το λόγο. Panie Κυρίες και κύριοι, για μας αποτελεί ιδιαίτερη ευχαρίστηση το γεγονός ότι μας καλέσατε σήμερα στην συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Για μας αποτελεί τη βασική ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις θέσεις της Πολωνικής Προεδρίας, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τον βασικό συνεργάτη του Συμβουλίου, και τρέφουμε απόλυτη συνείδηση κυρίες και κύριοι ότι οι επαφές με το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι επαναληπτικές, τακτικές και κυρίως στενές. Διότι έχουμε μια μεγάλη πορεία μπροστά μας αυτό το εξάμεινο και χωρίς εσάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλη αυτή η πορεία που έχουμε προβλέψει είναι σχεδόν αδύνατο να, να συνεχιστεί. Πρόκειται για μια... Είμαστε μια χώρα που πριν από 31 χρόνια μόλις πάλευε για την ελευθερία της. Πριν από 30 χρόνια βγήκαν τα τάξ στους δρόμους της Πολωνίας. Πριν από 30 χρόνια φυλακίστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είμαστε μια χώρα που εδώ και 22 χρόνια ξεκίνησε τις αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη. Πριν από 17 χρόνια μας υποδεχτήκατε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και πριν από 4 χρόνια μας επιτρέψατε να μπούμε σε αυτήν την κοινή Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Και υπ' αυτήν την έννοια δεν ε, θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι όταν ατενίζουμε από την Πολωνία την κοινή μας Ευρώπη, οι αξίες αποτελούν το θεμέλιο για μας. Γι' αυτό θέλαμε εμείς να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις αξίες για τις αξίες που προασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνες τις αξίες που είναι θεμελιώδεις και που αποτελούν φάρο. Για μας η λέξη αλληλεγγύη είναι μια σχεδόν ιερή λέξη, διότι αν δεν υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη πριν από 30 χρόνια, δεν θα είχατε υποδεχθεί εσείς τους πρόσφυγες από την Πολωνία μετά το πραξικόπημα εάν δεν είχαμε αλληλεγγύη πριν από 22 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε προσεγγίσει αυτή τη νέα το νέο δημοκρατικό σύστημα και χωρίς αλληλεγγύη δεν θα είχατε υποδεχθεί ένα γείτονα τόσο φτωχό στην οικογενειακή οικογένεια. Γνωρίζουμε καλά στο πετσί μας τι είναι η αλληλεγγύη και το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι το φυσικό, είναι κάτι που το ζήσαμε στο πετσί μας. Αυτό το οποίο εγώ ε, ε, θέλω να σας αναφέρω για την κοινή μας προσπάθεια στους επόμενους έξι μήνες είναι το εξής. Πρώτον ευχαριστήσω την Ουγγαρία η οποία εργάστηκε σκληρά και μας άφησε ορισμένα θέματα αρκετά προχωρημένα έστω και αν ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν. Εμείς Κατά συνέπεια θα ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία ξεκίνησε η Ουγγρική Προεδρία. Μεταξύ των βασικών θεμάτων θέλουμε να προωθήσουμε το θέμα του κοινού ευρωπαϊκού ασύλου που είναι ένα από τα πιο ισχυρά θέματα της Προεδρίας μας. Έχει προχωρήσει ιδιαίτερα το ζήτημα αυτό και σε λίγο καιρό θα μεταφραστεί σε εφαρμοστική οδηγία και όχι μόνο σε διαδικαστική οδηγία. Εμείς από τη μεριά μας, από την Πολωνική Προεδρία θέλουμε να προχωρήσουμε επίσης τις οδηγίες στην οδηγία υποδοχής και στην οδηγία διαδικασίας. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης όρισε ένα χρονοδιάγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο στα τέλη της επόμενης χρονιάς για να εφαρμόσουμε όλο αυτό το σύστημα. Ε, εμείς ε, σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε την πέμπτη ταχύτητα για να μπορέσουμε να τρέξουμε όσο πρέπει και να ολοκληρώσουμε τα θέματα αυτά. Γι' αυτό τις πρώτες ημέρες, ε, αυτές τις πρώτες μέρες του Ιουλίου οργανώνουμε αυτήν την συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για να εργαστούμε για την οδηγία υποδοχής και διαδικασίας. Τον Ιούλιο θα γίνουν δύο συνεδριάσεις και τον Σεπτέμβριο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν μιλάμε για το κοινό σύστημα ασύλου, θα πρέπει να μιλήσουμε για την Eurodap και το Δουβλίνο 3. Είμαστε, γνωρίζουμε όλοι τις πολεμικές που υφίστανται γύρω από τα θέματα αυτά. Αλλά είμαστε πεπισμένοι κυρίες και κύριοι ότι αναζητώντας έναν συμβιβασμό θα καταλήξουμε κατά τους επόμενους μήνες όλα τα έγγραφα να μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε. Θεωρούμε ότι είναι ένας ε, εφικτός στόχος. Το επόμενο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι η παράνομη μετανάστευση. τα κράτη-μέλη να υποδέχονται εποχιακούς μετανάστες ή εργαζόμενους αποσπασμένους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια οδηγία για την ενιαία άδεια και παραμονής. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν προχωρήσει. Αλλά απέχουμε αρκετά από την τελική λύση. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη θετική σας συνεργασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και τη σωστή λύση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει σε όλους μας. Όχι μόνο η δουλειά στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, αλλά και η δουλειά σε όλα, ε, σε όλα, τα επίπεδα, στα κοινά θέματα που μας καίνε όλους και αποτελούν στόχο και για τα κράτη-μέλη αλλά και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και για τις τρίτες χώρες που βρίσκονται στον περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οποίων η κατάσταση είναι άσχημη. και που η αστάθεια αυτών των χωρών επηρεάζει τα εσωτερικά της Ένωσης. Θέλουμε να υπάρξει μια αλλαγή, μια συζήτηση μάλλον ε, γύρω από τα σύνορα. Ξέρετε ότι η Πολωνία έχει ένα εξωτερικό σύνορο, έχουμε γείτονε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουμε καλά ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε με τους γειτόνους μας κοινά ε, ε, συνοριακή συνεργασία. Αυτό όμως χρειάζεται βάσεις και σε τεχνικό επίπεδο και σε διαπραγμάτευση. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι να καλέσουμε όλες αυτές τις ε, υπηρεσίες να μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί μας στα κοινά σύνορα. Μέχρι σήμερα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Και θα θέλαμε να ε, συζητήσουμε τις λύσεις των μεν και των δε. Θέλω, όταν μιλάμε για σύνορα θέλω να μιλήσω για τα ευφύη σύνορα. Σίγουρα στα σύνορα λείπει προσωπικό, λείπει κόσμος. Αλλά ε, χρειάζονται όμως ε, και άλλου είδους μέσα. Τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να είναι σύνορα τα οποία φρουρούνται καλά να μπορούμε ναι με να καλωσορίζουμε όσους μας έρχονται από τρίτες χώρες αλλά μπαίνουν παράνομα από αυτά, τα, σύνορα. Θέλουμε λοιπόν σύνορα σωστά φυλαγμένα. Όταν μιλάμε για τη ζώνη Schengen. Είναι σαφές. ότι στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική η κατάσταση είναι δύσκολη και για μας αποτελεί ένα τεστ. Γιατί σας το λέω. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε μια κατάσταση κρίσης, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και πώς μπορούμε να φυλάξουμε τα εσωτερικά μας σύνορα. Αυτό χρειάζεται μια τεράστια αναλυτική εργασία και μετά χρειάζεται και μια θεώρηση ε, ε, για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μηχανισμούς μπορούμε εμείς να, να, να αναλάβουμε για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη τη δυναμική του Frontex αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα συζητήσουμε η μεν και η δε όπως και το, να δούμε την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Μιλήσαμε για διάφορες λύσεις. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε φιλόξενοι έναντι αυτών οι οποίοι ζουν ε, ε, επικίνδυνα, αντιμετωπίζουν κινδύνους σε τρίτες χώρες. Αλλά πρέπει να τους διαχωρίσουμε από εκείνους που θέλουν απλώς να ζήσουν καλύτερα. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ύφεση. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και αυτές οι συζητήσεις, αυτή τη φάση, είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν. Εμείς ε, μιλήσαμε για τη σημασία συνεργασίας με τους γειτόνους μας. Ένας γείτονας ε, που προσέχει τα σύνορά του υπηρετεί καλύτερα την Ευρώπη από ότι έναν γείτονα ο οποίος αγνοεί την ύπαρξη σύνορων και η κατάσταση τόσο στα νότια σύνορα όσο και στα ανατολικά είναι ακριβώς η ίδια. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους πλησιέστερους γειτόνους για να λειτουργήσουν καλά τα κρατικά θεσμικά όργανα, τα εσωτερικά όργανα ασφαλείας υπέρ της προάσπισης των συνόρων. Σε αυτή τη φάση της Προεδρίας μας ε, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα δράσης. Όταν μιλάμε για την Ισία, Αίγυπτο, Μαρόκο, μπορούμε να μιλήσουμε και για Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, δηλαδή και τους ανατολικούς γειτόνους όσον αφορά στο οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών πρέπει να μιλήσουμε και για τα, ε, ναρκωτικά σύνθεσης. Τις νέες χημικές ψυχότροπες ουσίες. τις οποίες διακινεί το οργανωμένο έγκλημα μεν, αλλά αποτελεί δε και μια τεράστια απειλή για την υγεία των νέων. Και πρέπει να προετοιμαστούμε ούτω ώστε να σταματήσει αυτή η προσφορά των συνθετικών ναρκωτικών. Αυτά τα ναρκωτικά απαγορεύονται σε ορισμένες χώρες αλλά στην πράξη βλέπουμε να κυκλοφορούν στο δρόμο. Τελευταίο, Βουλγαρία, Ρουμανία. Εμείς το Δεκέμβριο του 2006 τον περιμέναμε, τον, τον περιμέναμε με αγωνία όταν γκρεμίστηκαν τα πολωνικά σύνορα. Και είχαμε πανηγύρια στο δρόμο. Και αν πει κανεί σε κάποιον Πολωνό ότι ορίστε τώρα θα κλείσουμε τα σύνορα και δεν μπορεί να πηγαίνει ελεύθερα όπου θε, ε τότε θα θυμώσει. Γι' αυτό θα κάνουμε ότι μπορούμε ούτω ώστε το συντομότερο δυνατό και η Βουλγαρία και η Ρουμανία να μπουν στο Σέγγεν. Έχουν όλα τα τεχνικά, πληρούν όλα τα τεχνικά ζητούμενα, οπότε θα πρέπει να μπουν στην οικογένεια το συντομότερο, το PNR τώρα. Γνωρίζετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα ολοκλήρωσης των συνομιλιών με, την, με τις Ηνωμένες Αυστραλία, Καναδά. Πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να διαπραγματευτούμε την τελική λύση και να βρούμε κοινές λύσεις αποδεκτές από όλους που να μας εγγυώνται επίσης την γρήγορη πληροφόρηση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Υπουργέ. Μείνατε και μέσα στα χρονικά σας ε, περιθώρια. Έχουμε προβλέψει μια μισή ώρα για, την ε, παρουσίαση και των, ε, για τις παρουσιάσεις και των δύο υπουργών. Οπότε, αμέσως μετά μπορούμε να κάνουμε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ε, φακέλους που είναι σημαντικοί. να θυμάστε ότι πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα σας. Οπότε τώρα προτείνω να πάμε στον δεύτερο υπουργό και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση, να ακούσουμε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Κουβιατκόφσκι έχει το λόγο. you got the floor now. Έχετε το λόγο, Υπουργέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ελπίζω η παρουσίασή μου να είναι πιο εύκολη από το όνομά μου. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργό Μίλλερ ε, μίλησε πολύ για αξίες, τις οποίες ε, συνδέουμε με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η πλειοψηφία των δράσεων που έχουν αναλυφθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις αφορούν κυρίως ε, μέτρα και ποινές για την αντιμετώπιση σοβαρών αδικημάτων και αυτή η προσέγγιση ήταν και είναι απολύτως κατανοητή γιατί τα ανοιχτά σύνορα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για να ξεφεύγουν ή να διαφεύγουν τις δικαιοσύνης αλλά στην παρούσα φάση θα θέλαμε να αλλάξει κάπως αυτή η προσέγγιση. Και γι' αυτό σας δίνουμε σήμερα το γενικό μας όραμα και τις προτεραιότητες της ε, Πολωνικής Προεδρίας σε σχέση με τα θέματα ΔΕΗ στα πλαίσια της προστασίας των δικαιωμάτων ε, των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για το δρόμο που μας έχει ανοίξει στον τομέα αυτό, ώστε να κάνουμε κι εμείς καλύτερα τη δουλειά μας. Κατά τη διάρκεια της ε, δουλειάς που έγινε για τα νέα προγράμματα, προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε αυτή την ε, ισορροπία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την ασφάλεια και εξασφαλίζοντας τα ελάχιστα δικαιώματα για τους κατηγορούμενους και τους υπόπτους. Από την άλλη, είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε επαρκή δικαιώματα τα οποία θα γίνονται σεβαστά και για τα θύματα. Γιατί τα θύματα δεν μπορούν να θεωρούνται ως αντικείμενα στην όλη διαδικασία. Η δημιουργία κοινών και προβλεπόμενων εχεγγύων και εγγυήσεων στις ποινικέ διαδικασίες είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό και βεβαίω πρέπει να το έχουμε υπόψη. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή περίπου 12 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής σε χώρα διαφορετική της χώρας γέννησή του. Κάποιοι από αυτούς έρχονται σε επαφή με διαφορετικά, με ξένα δικαστικά συστήματα. Και ακριβώς εδώ είναι που πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας πώς λειτουργούμε στην πράξη και πώς μπορούμε τελικά να επηρεάσουμε τα πράγματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Σημαντικό επίσης είναι να ολοκληρωθεί η οδηγία για το ένταλμα ευρωπαϊκής προστασίας. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το εργαλείο, γιατί μπορούμε έτσι να βασιστούμε σε στατιστικά στοιχεία τα οποία δυστυχώ δεν πρέπει να μας κάνουν και πολύ υπερήφανου, γιατί τα στατιστικά που έχουμε έρχονται από την Πολωνία και το 2010 ο αριθμό των θυμάτων οικιακή βία στην Πολωνία έφτασε πάνω από τις 130.000 άτομα. 82.000 αυτών ήταν γυναίκες και περίπου 40.000 ήταν παιδιά. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ασφαλείς στην Ευρώπη. Θυμηθείτε ότι τα σύνορα δεν είναι εμπόδιο και δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο ούτε για τους ε, θύτες ούτε για τα θύματα. Κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας θα ξεκινήσουμε την ε, δουλειά στις ομάδες εργασίας, στις εργασίας για, την, για το σχέδιο οδηγίας για την ε, καθιέρωση ελάχιστων προτύπων σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων ε, από αδικήματα. Και το πιο σημαντικό στο πλαίσιο αυτό είναι τα πιο ευαίσθητα, τα πιο ευάλωτα θύματα, όπως άτομα που είναι θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, εμπορίας ανθρώπων ή παιδιά. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε αρκετή πρόοδο ως προς αυτό τους επόμενους 6 μήνες. Και πέραν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος θα το συζητήσουμε αυτό και σε μια άτυπη συνάντηση τον το, με τους G8 που θα γίνει στο Σόμποτ και επίσης θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που γίνεται για τη σχετική οδηγία. Επίσης, ε, έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε την δουλειά στα πλαίσια του δικού χάρτη που έχει υιοθετηθεί, ο οποίος έχει στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Σημαντικό επίση είναι το γεγονό ότι η δουλειά που έχει γίνει για το σχέδιο οδηγία για το δικαίωμα σε ενημέρωση στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών ε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και επίση ζωτική σημασία είναι η συνεργασία η δική μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εσά, ε, κατά τι πρώτε μέρε που αναλάβαμε την ε, Προεδρία έχουμε ήδη ξεκινήσει εντατική δουλειά σε συνεργασία με εσάς, με το Κοινοβούλιο και σήμερα έγινε άλλη μία σύνοδος τριμερούς διαλόγου η οποία ελπίζουμε ότι θα μας φέρει πιο κοντά ακόμα στην εξέβρεση μιας λύσης που να είναι αποδεκτή από όλους. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά σας ως προς αυτό. Το σημαντικό επίσης για μας είναι το σχέδιο οδηγίας για την ε, πρόσβαση σε δικηγόρο στις ποινικέ διαδικασίες. Το να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα αυτό στην πιο πρώιμη δυνατή φάση της ε, ποινική διαδικασίας είναι, είναι σημείο κλειδί ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει και δίκαιη δίκη. Κατανοούμε βεβαίως ότι αυτό είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που μάλλον θα είναι και το πιο δύσκολο να συμφωνηθεί από όλον τον οδικό χάρτη. Γιατί ε, άπτεται πολύ σημαντικών πτυχών ε, των εθνικών δικαστικών συστημάτων. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι επικοδομητική η συνεργασία μας και θα καταλήξουμε τελικά σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να τελειώσουμε τη δουλειά λοιπόν που γίνεται ως προς αυτό, έχει ήδη γίνει αρκετή πρόοδος κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και αναφέρομαι κυρίως στον, στην εξασφάλιση των πολιτών μας σε ό,τι αφορά νέου τύπου επιθέσεις όπως οι κυβερνοεπιθέσεις. Το Συμβούλιο τον Ιούνιο υιοθέτησε μια γενική απόφαση, μια συμφωνία μάλλον, ε, για μια οδηγία που θα αφορά τις επιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής. Και θεωρούμε ότι ε, από κοινού μέσα με το Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να έχουμε αρκετέ ε, επαφέ στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου, έτσι ώστε στο τέλο του χρόνου να δείξουμε συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα τη δουλειά μα. Και επίση κάτι άλλο που άφησα για το τέλος, αλλά νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό. είναι η φόβη που έχω. Πιστεύω πως ε, το Κοινοβούλιο, όπως και εμείς, είναι αφοσιωμένο στο να αντιμετωπίσουμε την ε, παιδική εκμετάλλευση. Χαίρομαι που τα αποτελέσματα του, των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας οδήγησαν σε έναν πολύ ουσιώδη συμβιβασμό και τώρα ως ε, Προεδρία και προς όφελος των θυμάτων βεβαίως ελπίζουμε να υπάρξει μια λύση που θα είναι λίγο πιο ευρεία. Υπάρχουν ε, κάποια ενισχυτικά σημάδια ακόμη ε, που έρχονται προς το Συμβούλιο γιατί φαίνεται ότι αυτή η συμβαστική πρόταση μπορεί να απειλείται. λόγω των πινάκων ισοτιμίας, αλλά, αντιστοιχίας. Αλλά αυτό πραγματικά μας ανησυχεί πάρα πολύ και θα πρέπει να το δούμε. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου πως το πρόβλημα αυτό είναι οριζόντιας φύσης και δεν θα πρέπει να μπλοκάρει αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες όπως είναι η προστασία των παιδιών ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που εκπροσωπώ μία από τις πρώτες ε, προεδρίες που συνεργάζεται εδώ με εσάς, με το Κοινοβούλιο, στα θέματα ποινικών διαδικασιών ώστε να υπάρξουν νέοι κανόνες στα πλαίσια της συναπόφασης, όπου και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι ισότιμοι εταίροι. Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών θα μπορέσουμε να σας δείξουμε ότι αυτή η συνεργασία είναι ιδιαίτερος αποτελεσματική και είναι η κινητήριος δύναμη για την ε, εκπόνηση της περαιτέρω πολιτικής για τον τομέα της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ευαίσθητα τα θέματα που θέσατε και είναι ζητήματα που μας απασχολούν όλους, όλος ιδιαίτερο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι εκ μέρους της Επιτροπής ΛΥΠΕ θα συμμετάσχω στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Συστημάτων που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα στο Σόποτ, στην Πολωνία, στο πλαίσιο της Πολωνικής Προεδρίας. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. 23 αν μέτρησα καλά. Οπότε προτείνω την εξή διαδικασία. Πρώτον, πρώτα συντονιστέ. Κάθε πολιτική ομάδα θα λάβει το λόγο και στη συνέχεια θα ακούσουμε έναν πρώτο γύρο απαντήσεων και από τους δύο υπουργούς. Μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο με τους υπόλοιπους συναδέλφους και θα ήθελα να σας ζητήσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτά για να έχουμε αρκετό χρόνο. Αν υπερβείτε το χρόνο σας, θα χτυπάω το σφυράκι. Λοιπόν, αρχίζουμε με τους συντονιστές, όπως είπα. Ο κύριος Σόμπου θα έχει το λόγο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας και ε, εγώ θα κάνω μόνο μία ερώτηση. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Ε, ποια είναι τα σχέδια της Πολωνικής Προεδρίας σε σχέση με τη γενική προσέγγιση ε, με, τη μετανάστευση και στο πλαίσιο της ανατολικής πολιτικής γειτονία. Ευχαριστώ πολύ. Και ήσασταν και πάρα πολύ σύντομο. Σας ευχαριστώ διπλά λοιπόν. Για τους σοσιαλιστές, η κυρία Ζίπελ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την πορτογαλική διερμηνία, λέει ο κύριος Κοέλιο. Υπάρχει τρομερός θόρυβος και δεν μπορώ να ακούσω τίποτα. Ο πρόεδρος ε, ρωτά αν μπορεί να γίνει κάτι για την πορτογαλική προεδρία, ε, πορτογαλική ε, διερμηνία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μόνο τα πορτογαλικά έχουν πρόβλημα. Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ε, μπορώ να ακούσω ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά, λέει ο κύριος Κοέλιο, αλλά νομίζω ότι είναι απλώς τεχνικό το πρόβλημα. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος, ελπίζω να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Η κυρία Σίπελ για τους σοσιαδημοκράτες. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους υπουργού για την παρουσίασή τους. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες συζητήσει που κάνουμε, γιατί μιλούμε για βασικές αξίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αλληλεγγύη, και πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι αυτές τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας μόνο μαζί μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί πρέπει να φροντίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, αλλάξουμε τα πράγματα αλλά και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αλλάξουν κάπως οι συνθήκε, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν λέω ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα των ε, συνόρων και των ελέγχων στα σύνορα για την συνεργασία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ε, είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι οι νέοι έλεγχοι δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στο ότι η ε, εγκληματικότητα θα αντιμετωπιστεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται στενή συνεργασία με, το, με τα κράτη-μέλη και στα πλαίσια της, του, των δικαστικού τομέα αλλά και στα πλαίσια της αστυνομία. Πρέπει και τα εθνικά συστήματα να κάνουν κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να είμαστε τελικά αποτελεσματικοί στη δουλειά μας και να μην ε, αφήνουμε τους εγκληματίες να αλωνίζουν σε εισαγωγικά. Πάμε τώρα στους, ε, στα δεδομένα των ε, επιβατών των αερομεταφορών. Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις ε, για τι μεταφορέ αυτέ. και ελπίζω η Προεδρία να προχωρήσει τι διαπραγματεύσει που κάνει με, τις, ε, με την Αμερική, με τις ΗΠΑ. Τώρα για την πολιτική ασύλου και τη μετανάστευση είναι σημαντικό και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μελλοντικά στα κράτη-μέλη μα θα χρειαστούμε μετανάστευση έτσι ώστε, έτσι ώστε τώρα, μάλλον θα πρέπει τώρα να στείλουμε τα σωστά μηνύματα γιατί είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δυνατότητε, ευκαιρίε, ακόμη και για αυτού που ήδη είναι στα, στα κράτη-μέλη μας τώρα και ζουν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Aldi Group. Για την ομάδα των φιλελευθέρων, κυρία... Thank you, Minister. Βέμπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Μίλλερ και τον κύριο Κφιατκόφσκι για την παρουσίασή τους ανεξαρτήτως της γλώσσας που μιλούμε πολωνικά, ρουμανικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, μπορούμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα όταν ε, βασιζόμαστε στις ίδιες αρχές και στις ίδιες αξίες. Και πραγματικά εκτιμώ όλος ιδιαίτερος τα εισαγωγικά σας σχόλια επ' αυτού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης για όλα όσα είπατε για την ε, άποψη των Πολωνών για τη, για τη ζώνη Σέγγεν. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό ήταν ε, όταν ε, προσχωρήσατε στη ζώνη αυτή και θα ήταν πολύ δυσάρεστο να ε, αλλάξει αυτό. Στο περασμένο του ψήφισμα για το θέμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι θέλει να χτίσει πάνω στο κεκτημένο της Σέγγεν και δεν θέλει επιπλέον ελέγχους στα σύνορα. Θα ήθελα, κύριε Κφιατκόφσκι, ε, κύριε Υπουργέ, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι εύκολο ε, ε, για την πρόσβαση στο δικηγόρο και για την προστασία των θυμάτων. Δεν ξέρω πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί είναι γεγονός ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα της βίας κατά των γυναικών, τουλάχιστον για, την, ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και μιλώ για τη σχετική έκθεση. Και για τον Υπουργό Μίλλερ, προς τον Υπουργό Μίλλερ θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ με όλα όσα άκουσα για το άσυλο. Το θέμα είναι πώς βλέπετε το ότι πριν από δύο εβδομάδες η Γαλλία, η Αγγλία και η Γερμανία προέβησαν σε μία δήλωση που ήταν κατά κάποιο τρόπο μία δήλωση πολέμου. Εντάξει, ας μην το πω τόσο τραβηγμένα, αλλά ουσιαστικά αυτό λέει, αυτό που είπαν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε ένα σύστημα ασύλου, ότι πρέπει να παραμείνουμε με ε, το τρέχον status quo. Είναι μία άποψη με την οποία εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, Αντιθέτω μάλιστα, Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς έχετε σκοπό να εργαστείτε για την προστασία δεδομένων ε, και το PNR Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε ό,τι υφίσταται αυτή τη στιγμή ε, ό,τι υπάρχει στην σχετική συμφωνία να μην είναι ενάντια στη δική μας προστασία δεδομένων. Για τους πράσινους η κυρία Σαρζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο Πολωνούς Υπουργούς που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ καλό που έχουμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές τη δυνατότητα να ε, ανταλλάξουμε απόψεις. Κάποια μέλη της Επιτροπής μας θα μεταβούν στην Τινησία σήμερα το πρωί. Μας ενημέρωσαν για τον αριθμό των προσφύγων ε, αυτή τη στιγμή στην Τινησία και τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν, αντι... που έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα γιατί δεν μπορούν να γυρίσουν ε, στη χώρα τους. Από ό,τι κατάλαβα, οι Πολωνοί έχουν υποδεχθεί 16 χριστιανούς πρόσφυγες από την, ε, την Ισία. 16, 10 συν 6. Πολύ καλή αρχή, αλλά υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες από την Ερυθρέα, τον Τακφούρ, τον Λαφούρ, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, χώρες ε, στις οποίες δεν μπορεί να επιστρέψει κανείς και να μην ξεχνάμε και την ακτή του ελεφαντοστού. 800, 800 με 900 θέσεις έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στους ανθρώπους αυτούς, το ίμιση των οποίων ε, αφορούν ε, προ, πρόσφυγες που έχουν ήδη φτάσει σε ευρωπαϊκές ακτές και όχι στους πρόσφυγες ε, τους οποίους θα επισκεφθούμε στους διάφορους καταφλισμούς στο σύνορο με τη Λιβύη. Η Πολωνική Προεδρία μήπως βλέπει ευκαιρία καταρχάς αύξησης ε, του αριθμού ε, των ε, προσφύγων που θα υποδεχθεί πάνω από 16 εννοώ, όπως επίσης και να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του επαναπατρισμού της επαναπροώθησης που δίνει τη δυνατότητα που βοηθά τους την ίσιους πρόσφυγες. Το άλλο θέμα αφορά την νομική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για τη νομική βάση για το και εκτιμένο Σέγγεν. Η συνάδελφος Βέμπερ το ανέφερε ήδη την, ε, το ψήφισμα της περασμένης εβδομάδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει τουλάχιστον, επιμένει τουλάχιστον στο άρθρο 77 που μας δίνει συναπόφαση για τη Σέγγεν και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ορισμένα μέλη ε, στο Συμβούλιο που θέλουν να αλλάξουν τη νομική αυτή βάση και θέλουν ε, να απομακρύνουν τη δυνατότητα ε, συναπόφασης ε, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ένα ακόμη ερώτημα το οποίο κάπως θίξατε είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Πήγα προσφάτως στην Πολωνία μαζί με έναν Ολλανδό πολίτη για τον οποίο υπήρχε ένταλμα συλλήψεως αν δει κανεί τι στατιστικές για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι γεγονό ότι η χώρα σα υπερβαίνει όλες τις υπόλοιπες ε, χώρε τα κατά πολύ. Υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών σε σχέση με το τι αποτελεί έγκλημα και μάλιστα έγκλημα το οποίο μπορεί να έχει ω αποτέλεσμα αυτό το ένταλμα Συλλήψη. Υπάρχουν διαφορετικέ δυνατότητε κράτηση. Ο Ολλανδό συνάδελφο συνάδελφος έμεινε σε προδικαστική διαδικασία μόνο για δύο μέρες. Ε, δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του και οι εγκαταστάσεις κράτησης σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης είναι σε τέτοια κατάσταση που πραγματικά δεν είναι καθόλου ε, υγιεινό να υπάρξει ένταλμα σύλληψης για κανέναν αν πρόκειται να κρατηθεί σε, αυτά τα, σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Μήπως, ε, μήπως προβλέπετε μία αλλαγή για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Εγώ θα ήθελα να σας ε, καλέσω να το κάνετε και να δείτε και το θέμα της αναλογικότητας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΙΣΙΑΡΟ, ο κύριος Κύρκοπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ Ελπίζω η Πολωνική Προεδρία να είναι επιτυχής ε, και ακούγοντας τα σχόλια των δύο προσκεκλημένων ομιλητών μας ε, υπάρχουν ε, αρκετές, αρκετοί τομείς που χρήζουν προσοχής και που είναι πολύ σημαντικοί. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις σύντομες. Πρώτον, το θέμα το, των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ζώνης του Σέγγεν. Αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσαν οι προσκεκλημένοι μας να εμβαθύνουν λίγο σε αυτό, γιατί υπάρχει, έχει ακουστεί ότι θα αλλάξουν τα κριτήρια ή ότι θα υπάρξουν κάποιοι ε, συνοριακοί έλεγχοι σε μερικές περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ε, όταν ο Πρωθυπουργός σας ε, Τάσκ είπε στην... Ε, ε, αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα και στο Στρασβούργο και μίλησε για το Ευρωπαϊκό Κοινό ε, Σύστημα Ασύλου. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι μιλάμε για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες του 1951 που μέχρι τώρα μας έχει δώσει τα κριτήρια χορήγηση ασύλου. Θα ήθελα επίση να ακούσω τα σχόλιά σα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, για τα ε, συστήματα πληροφορικής Στάλιν, Στράσβουργκ ε, και uh, και σε μία πόλη της Αυστρίας θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για την ενδεχόμενη δημιουργία ε, ενός ε, οργανισμού που θα εντοπίζει τους ε, τρομοκράτες. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, για το θέμα των του PNR. Φτάνουμε ε, στα 10 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ε, έγιναν και τρομοκρατικές επιθέσεις στο Λονδίνο. Ε, πώς θα αποτελέσουν αυτά προτεραιότητες προκειμένου να στοχεύσουμε ειδικότερα το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ. E, Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Άρνστ για την ΚΟΕ. E. Ευχαριστώ. Ε, ό,τι καλύτερο στην ε, Προεδρία σας. Ε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ελπίζουμε να έχουμε καλή συνεργασία. Ένα σημείο θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο είναι η Schengen. Ξέρετε ότι στο Κοινοβούλιο στις διάφορες συζητήσεις που γίνονται υπάρχει μεγάλη κριτική από πολλούς ευρωβουλευτές για την επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων και συνέχεια λέγεται ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου διαφανή ως προς αυτό. Η Σέγγεν αποτελούσε ένα σύμβολο για την Ευρώπη και δεν μπορούμε να την, κατα... να την καταστρέψουμε και μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, σε εξαιρέσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν ίσως κάποιες ρυθμίσεις για τέτοιους ελέγχους. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, Έχουμε Έχετε κάποια κάποιο σχέδιο. Επίσης είπατε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ανοιχτή για αυτούς που για ε, χρηματικούς λόγους έρχονται εδώ. Αυτό τι σημαίνει όμως. Μιλούμε για εργάτες από, το Μάλι, από την Ιγυρία, από τον Νίγηρα, από... Εντάξει, από το Νίγηρα όχι τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ε, Μιλούμε για τέτοιους ανθρώπους που έχουν εργαστεί σε κάποιες χώρες και τώρα λόγω των εμφυλίων πολέμων που γίνονται στη χώρα τους ε, φεύγουν. Αλλά θέλουν να, βολε... θέλουν να δουλέψουν, δεν θέλουν να, γίνουν, ε, να ζητήσουν άσυλο. Τι θα κάνετε με αυτό. Επίσης, είναι σωστό να υπάρχει χρονικά περιορισμένη προστασία αυτών των ατόμων ώστε να τους δίνεται η πιθανότητα να βρούνε ε, δουλειά στην Ευρώπη. Και επίσης, ε, θα μπορούσαν ίσως αργότερα να επιστρέψουν στη χώρα τους. Βλέπετε καθόλου ανάγκη αλλαγής των ε, συστημάτων ασύλου. Έχετε κάποιο, κάποιο σχέδιο προς αυτό. Και άλλο ένα σημείο, προστασία των δεδομένων. Υπάρχει η οδηγία η οποία τώρα την χάνει μελέτη επεξεργασίας ε, εγώ δεν ήμουν σε όλη την παρουσίασή σας ε, στο, στην αίθουσα, αλλά ίσως να είπατε κάτι. Αλλά αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κατά τη διάρκεια της προεδρία σας, τι θέλετε να επιτύχετε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, τι θέλετε δηλαδή να προχωρήσετε, να προωθήσετε, ώστε να υπάρξουν και κάποιε αλλαγέ στην οδηγία. Και τελευταίο σημείο. Ένα μεγάλο θέμα σε πολλέ συνεδριάσει αυτή τη επιτροπή ήταν το θέμα της μη διακριτικής μεταχείρισης και η αναγκαία προστασία των ομοφιλοφίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνική Προεδρία θα δώσει μια όθηση προς τα μπρος στο θέμα αυτό, ώστε να υπάρχει μια εξίσωση των ατόμων αυτών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων τώρα με την ίδια σειρά. Αλλά ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια δεύτερη σειρά ερωτήσεων, οπότε θα πρότεινα να μην μας διαφεύγει, να μην μας διαφέρει και το θέμα του χρόνου. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να απαντήσετε επί της ουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, μην ανησυχείτε, Πρόεδρε, έχω το ρολόι μπροστά μου. Μιλήσαμε για την ε, ανατολική συνεργασία και για τη συνεργασία στα σύνορα. Απαντώ. Οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Αν θέλουμε κατά συνέπεια να παλέψουμε κατά της εγκληματικότητας πρέπει να συνεργαστούμε με τις φιλικές προς χώρες έχοντας πάντα συνείδηση ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, η αστυνομική συνεργασία για να μπορέσουμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Πρέπει όμως να συμμεριστούμε ό,τι κατέχουμε ως know-how Πρόκειται για μία μακρόχρονη διαδικασία. Αλλά όταν μιλάμε για συνεργασία, μιλάμε για κοινέ δράσεις προς το καλό όλων και των μεν και των δε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να έχουμε υπόψη μας ότι μπορούν να μας προστατεύσουν, ότι μόνο έτσι μπορούμε να προστατευτούμε από το οργανωμένο έγκλημα για την μετανάστευση τώρα. Αλλά λάβουμε υπόψη τις αλλαγές στην Βόρειο Αφρική. Να, από τη Λιβύη έφυγαν 900.000 άτομα. Μα κανένας δεν του πέρασε από τον νου όμως αυτά τα 900.000 άτομα τα φέρει στην Ευρώπη. Πρέπει εμείς να προστατεύσουμε αυτές τις 900.000 στη χώρα τους, όχι να τους φέρουμε στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ σύνθετη όμως αντίληψη αυτή. Δεν είναι μόνο μια, μια όψη της πολιτικής μετανάστευσης. βρισκόμαστε σε μία περίοδο κρίσης και η βοήθειά μας πρέπει να προσεγγίζει την ίδια την Αφρική, όχι μόνο την Λαμπεντούζα. Ε, κάποιος έρχεται με ένα καΐκι, με μια ε, σχεδία στην Ευρώπη ε, πρέπει να βοηθηθεί όχι πια στην Ιταλία, στη χώρα του για να μην χρειαστεί να φύγει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την, το πρόβλημα της μετανάστευσης συγκεντρωμένο μόνο σε ένα νησί. Είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο πολύπλοκο πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την οικονομική βοήθεια. Εάν εμείς μιλάμε για πολιτική μετανάστευσης, Δείτε τι γίνεται, είχαμε αυτές τις 16 οικογένειες που ήρθαν στην Πολωνία. Και η Πολωνία έκανε μία ε, πρόσκληση και δέστε στη Μάλτα, ας πούμε, πρόσφυγες από τη Λιβύη. Κανένας δεν δέχτηκε την πολωνική πρόσκληση. Διότι φυσικά η Πολωνία δεν εντάσσεται στα μεταναστευτικά σχέδια, δεν είναι μία ένας θελκτικός προορισμός, αλλού θέλανε να πάνε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε η μεταναστευτική και η πολιτική της Ευρώπης να είναι ενιαία Πρέπει να έχουμε μία ενιαία φωνή και να μπορούμε να, μοιράζουμε αυτό το βάρος. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι στη Σουηδία πάνε 200.000 μετανάστες το χρόνο ενώ στην Πολωνία μόνο 10.000 το χρόνο. Πρέπει λοιπόν αυτό το βάρος να δούμε πώς θα το μοιράσουμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερα ποσοστά αιτήσεων ασύλου και που δίνεται αυτό το άσυλο τελικά. Ενώ σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρει κανείς το άσυλο. Πρέπει να εφαρμόσουμε τους ενιαίους όρους ασύλου και μετανάστευση σε ένα κοινό πακέτο. Και πρέπει να ρυθμιστεί πια αυτός ο μηχανισμός. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί αυτός ο μηχανισμός. Μη με παρερμηνεύετε, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στην τωρινή κατάσταση. Προηγουμένως ε, κάποιος είπε αν αυτό είναι συμβατό με τη σύμβαση της Γενέβης. Μα φυσικά και σε μερικές μέρες θα έχουμε τα 60 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης της Γενέβης. Το 51 υπογράφτηκε και αποτέλεσε μοντέλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν στον Ταμπέρε έγιναν τα πρώτα βήματα για την προστασία των προσφύγων που φεύγουν από τις χώρες τους για να έρθουν στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος με ρώτησε για το Σέγγεν. Ο κύριος Κύρχοπ νομίζω με ρώτησε. Μα σας το είπα και πριν. Η εσωτερική και η εξωτερική κατάσταση θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μία εις ανάλυση της κατάστασης. οι λύσει που έχουμε μπροστά μας είναι λύσει που δεν είναι κατάλληλε για τη νέα εποχή που περνάμε για το 2011. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη θέση του. Διότι υπάρχει ένα σαφές μήνυμα ότι η ελευθερία διακίνησης μέσα στο Σέγγεν είναι πολύ σημαντική. Αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν βασικό δίχτυ των όλων όσων θα συζητήσουμε. Υπάρχουν όμως χώρες όπου ολοκληρώνονται ορισμένες δράσεις που αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει αν είναι συμβατές ή όχι με το κοινοτικό δίκαιο και αν παραβιάζουν το δίκαιο τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για το Συμβούλιο ΔΕΗ στο Σόμποτ περιμένουμε τους υπουργούς εσωτερικών υποθέσεων να δηλώσουν ε, σαφώς ποιες είναι οι προθέσεις τους για όλα τα θέματα που αφορούν τη μετανασύλου για την περιοχή της Σέγγεν και όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της από ε, εδώ και χρόνια. Βεβαίω ε, τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, κατακαιρματισμένα. Δεν μπορεί η χώρα Α να δρά διαφορετικά από τη χώρα Β, γιατί αλλιώ δεν ε, δρούμε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να έχουμε έτσι ημίμετρα. Δεν είναι, αυτός, δεν είναι αυτή η κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συνοριακούς ελέγχους. Πρώτον, θέλουμε τα σύνορά μας να είναι φιλικά προς όλους όσους θέλουν να διέρθουν των συνόρων. Υπάρχουν ε, άνθρωποι που έρχονται συχνά ε, στην, ε, στις χώρες μας και που δεν έχουν καμία πρόθεση να διαπράξουν κάποιο έγκλημα ή κάποιο αδίκημα. Οπότε πρέπει να διευκολύνουμε την ε, διέλευση αυτών. Αλλά βεβαίως αυτό πρέπει να το δούμε πάντα αναλογικά γιατί υπάρχουν πολλές φορές και δυνατότητες ε, να υπάρξει κατάχρηση αυτών των ε, διαδικασιών στα σύνορα. Θα δούμε αν ας πούμε, μπορούμε να, υπάρξει, να δώσουμε δυνατότητα στους συνοριοφύλακες να ελέγχουν ε, όσους περνούν τα σύνορα και αν μπορούμε κάποιον να τον διώξουμε εφόσον έχει λήξει η θεώρησή του. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε όμως πόσες περιπτώσεις ε, τέτοιας παράνομης παραμονής έχουμε, μετά τη λήξη δηλαδή των θεωρήσεων. Ε, ξέρω ότι ε, τελειώνει ο χρόνος μου, αλλά έχω να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει, υπάρχουν δύο συστήματα τα οποία έχουν προχωράσει σε πάρα πολύ. Το σύστημα των θεωρήσεων, το οποίο ήδη θα μας βοηθήσει να εκδώσουμε από το Σεπτέμβρη και μετά θεωρήσεις ε, για τα άτομα που έρχονται στην Ευρώπη από τις χώρες της Βορειοφρικής και της Μέσης Ανατολής. Και το άλλο σύστημα είναι το σύστημα ΣΥΣ2 το οποίο μπορεί να αρνηθεί την είσοδο κάποιων ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μπορεί να καταγράψει ποιε ήταν οι δράσει κάποιων ατόμων όταν φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συστήματα αυτά λοιπόν είναι λειτουργικά. Αλλά το δεύτερο σύστημα εξακολουθεί να, το δεύτερο σύστημα ήδη εξακολουθεί να ε, ήδη εφαρμόζεται. Οπότε όταν μιλούμε για τέτοια συστήματα και για υπηρεσίε πληροφορική, θα πρέπει να μιλούμε και για καλέ και για κακέ εμπειρίε. και θα πρέπει να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε με τον καταλληλότερο τρόπο τα χρήματα των φορολογούμενων μας. Τώρα, ο Υπουργό Κβιατκόφσκι, κανεί δεν θέλει να είναι γενή απέναντι στου υπουργού προφανώ. Ε, Απλώ επειδή είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο, ε, θα σα ζητήσω να είσαστε κι εσεί όσο σύντομο μπορείτε να είστε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εγκαρδίως ε, τους συναδέλφους ε, για τις ερωτήσεις τους και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα την κυρία Βέμπερ, γιατί για την οικογενειακή βία ενδιαφέρομαι πάρα πολύ. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μία από τις πρώτες αποφάσεις μου αφορούσε αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα. Ε, μάλιστα ε, υπάρχει πλέον ε, ένας συντονιστής ε, που ασχολείται ειδικότερα με αυτά τα θέματα, αναλύει την νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για εργαστήρια και σεμινάρια που αφορούν αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και ορισμένες αλλαγές που έγιναν με αποτέλεσμα την μείωση του φαινομένου αυτού στην Πολωνία. Γι' αυτό ακριβώς Δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Η κυρία Σαρτζεντίνη έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Θα ήθελα να να αναφερθώ σε αυτό το θέμα λίγο παραπάνω. Είναι πραγματικά ένα κόσμημα της, ε, των μέσων ε, ε, ποινική συνεργασίας που έχουμε και αυτό βέβαια γιατί ήταν πολύ μακρόχρονη η διαδικασία έκδοσης και πολύ φορτωμένη. Είμαστε πράγματι μια χώρα που εκδίδει πάρα πολλά τέτοια εντάλματα και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως ε, δεν θα ήταν ε, σωστό να πει κανείς ότι το ένταλμα αυτό συλλήψεως αφορά μόνο σοβαρά αδικήματα. Υπάρχει μια απόφαση πλαίσιο που υποκαθιστά την ε, διαδικασία έκδοσης και είναι και έχει ακριβώ ε, το ίδιο πεδίο εφαρμογή ε, με την διαδικασία έκδοση. Οπότε, πρόκειται για δικήματα για τα οποία μπορεί κανείς να φυλακιστεί για ένα χρόνο ή και παραπάνω. Επομένως, ε, δεν υπάρχει περιορισμός στην έκδοση εντάλματος, τέτοιου εντάλματος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αποδυναμώνεται έχουμε λάβει επαρκή, έχουμε αναλάβει επαρκή δράση ε, βάσει των αποφάσεων του ε, Συμβουλίου και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πέρσι ένα εγχειρίδιο, το εγχειρίδιο διαδικασιών άλλαξε, τροποποιήθηκε από το ε, Συμβούλιο και θα δούμε σύντομα τα αποτελέσματα της, των, των αλλαγών αυτών, τροποποιήσεων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για κάποια μέτρα άλλα στην Πολωνία. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι για ένα χρόνο μόνο, αν συγκρίνουμε τα δεδομένα για το 2010 για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε το 2010 με το 2009, ο αριθμός των ε, εντάλματων ε, ε, μειώθηκε κατά 25% από 4.844 το 2009 σε επίπεδο σε 3.750 για το 2010. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των Πολωνών που ζουν εκτός Πολωνίας είναι αρκετά σημαντικός. Είμαστε βέβαια ανοιχτοί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το μέλλον του μέσου αυτού βάσει συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων και ε, δικαιολογημένων επιχειρημάτων. Προφανώς, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα, υπάρχει ένα περιθώριο καταχρήσεων, αλλά ακόμα και όταν υπάρχουν δυσανάλογα μέτρα, δεν θα έπρεπε να μειώνεται η εμπιστοσύνη μας σε ένα μέσο το οποίο λειτουργεί καλά και που είναι επιτυχές. Προφανώς η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται σε κάποιες αδυναμίες του συστήματος ε, και αναφέρει το δικαίωμα σε ε, ε, νομικές συμβουλές σε δικηγόρους. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, μέχρι τις 4.30 έχουμε χρόνο δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα καθυστερήσουμε λίγο να αρχίσουμε την ψηφοφορία μας, αλλά έχουμε ακόμη 18 μιλητές. Είχα πει δύο λεπτά ο καθένας. Ε, κάποιοι τα κατάφεραν με τα δύο λεπτά, κάποιοι σχεδόν τα κατάφεραν, αλλά πραγματικά ε, τώρα η μόνη επιλογή που έχουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερους είναι να έχει ο καθένας ένα λεπτό στη διάθεσή του, διαφορετικά δεν ε, θα μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο. Άρα, προτείνω. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας ζητήσω ότι έχετε στη διάθεσή σας ένα λεπτό. Ένα λεπτό το πολύ. Πρώτος, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και πολλές ευχές για τους ε, δύο υπουργούς. Εχθές ε, μια ισπανική φρεγάδα ε, μάζεψε στα νυχτά στη Μεσόγειο 100 άτομα και πήγε στο και προσεγγίζει στο λιμάνι της Σύρτης όπου αρνούνται να τους παραλάβουν οι Τινήσοι. Τι θα τους κάνουμε, τους έχουμε στη μέση της Μεσογείου σε ένα πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο. Τι θα τους κάνουμε, η Μάλτα θα πει δεν τους θέλω, η Ιταλία θα βρει κάτι άλλο να πει, τι θα πει το Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα για το άσυλο, Eurodac, Δουβλίνο 3 κλπ. Σύμφωνα με την πολιτική της Χάγης έπρεπε να είχαμε το 2010 μια πολιτική ασύλου. Και εσείς μας λέτε ότι σαν την καλή χαρά το 2012 θα την έχουμε αυτή την πολιτική. Λοιπόν, ποιες είναι οι δυσκολίες αλήθεια. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω λιγότερο από ένα λεπτό. Να ευχαριστήσω τους υπουργούς που ήρθαν στη συνεδρίαση και πάνω από όλα να τους ευχαριστήσω για το άνοιγμα τους προς το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να θέσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν τον έφερε κανείς στο πρόγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας ούτε και οι υπουργοί το ανέφεραν και αφορά πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Αναφέρομαι εδώ στην αμοιβαιότητα των θεωρήσεων πέντε κρατών μελών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αυστραλίας και του Καναδά και μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών χωρών λοιπόν υπάρχει και η Πολωνία. Κάνετε κάτι για να καταργηθούν οι βίζες με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά. Κάτι είπε στην Κολωνία ο πρόεδρος Ομπάμα, αν δεν κάνω λάθος. Η κυρία Αλφάνο για ένα λεπτό βέβαια πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, άκουσα από τους ε, Πολωνούς υπουργούς ότι σκέφτονται ότι δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα της τρομοκρατίας. Αλλά πέρα από τα θύματα της τρομοκρατίας έχουμε και τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος που είναι πάρα πολλά. Και επίσης αναφέρθηκαν και στην καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών Θεωρώ εξοφλημένο ότι η προσοχή σας θα στραφεί και κατά των παραγωγών και διακινητών ναρκωτικών. Σας τα ρωτώ αυτά γιατί εγώ είμαι συγγήτρια της έκθεσης για το οργανωμένο έγκλημα που θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο υπό την Προεδρία σας στη Μήνη Ολομέλεια. Η Ουγγρική Προεδρία έκανε πολλά πράγματα σε αυτό το μέτωπο. Εσείς το θεωρείτε προτεραιότητα και πώς θα το αντιμετωπίσετε. 56 δευτερόλεπτα, Πρόεδρε, μόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σημεία ήθελα να θίξω. Το ένα είναι το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης στις ποινικέ διαδικασίες Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η Προεδρία, δηλαδή η Πολωνική, να συνεχίσει να προχωρά στο δρόμο της κατάρτισης των ελάχιστων προτύπων, ανάλογα και στα πλαίσια βέβαια του οδικού χάρτη, ε, ώστε να ικανοποιήσει και λίγο το Κοινοβούλιο ε, το οποίο προσπαθεί τα ε, πρότυπα τα οποία είχαν παραβλεφθεί λίγο τα τελευταία χρόνια να τα επαναφέρει. Πρέπει λοιπόν και τα κρατημέλη να συμφωνήσουν, είναι σημαντικό αυτό. Ένα δεύτερο σημείο ε, είναι ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι είμαι μόνος, ε, το πρόβλημα της, ε, του οικονομικού εγκλήματος, ας πούμε αντιμετώπιση του ξεπλήματος σε μαύρου χρήματος και άλλων μορφών, να τα βάλουμε στον πυρήνα της συζήτησής μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίω και σε θέματα όπω η ε, τρομοκρατία και η αντιμετώπιση τη. Ε, πρέπει να θέσουμε λοιπόν σωστέ ε, προτεραιότητε ω προ αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κλέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι η Πολωνική Προεδρία θα συνειδητοποιήσει πλήρως ότι βρισκόμαστε σε μια υπαρξιακή κρίση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλούμε απλώς για προβλήματα στην Ευρωζώνη, μιλούμε και για προβλήματα σε με την ελευθερία κίνηση των πολιτών ή των ατόμων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η συμφωνία της Σέγγεν, αλλά είναι, ε, εφαρμόζεται μερικώς. Δεν υπάρχουν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, αλλά τι γίνεται με τα εξωτερικά σύνορα. Εκεί είναι έτσι σαν δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τίποτα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε ας πούμε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η σοβαρότητα της κατάστασης πραγματικά είναι ιδιαίτερη και ελπίζω η Πολωνική Προεδρία να τη γνωρίζει. Πριν από κάποιες εβδομάδες έγινε μια, συμφωνία στην τελευταία σύνοδο και υπόθηκε ότι θα υπάρξει συμφωνία με τις τρίτες χώρες για να αντιμετωπιστεί η παρανομή μετανάστευση. Πρόσφατα υπόθηκε αυτό αυτή η συμφωνία όμως τι θα περιλαμβάνει. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ως προς αυτό. Η Προεδρία θα προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο. Επίσης, με τα εξωτερικά σύνορα τι γίνεται. Αυτή είναι η δική μου ανησυχία. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ο κύριος Κοέλιο για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους Υπουργούς για την παρουσία τους και για τις δηλώσεις που έκαναν. Και κυρίως για αυτό το οποίο είπαν σχετικά με το Σέγγεν. Ξεκίνησαν έγκαιρα να ετοιμάζουν αυτή την Προεδρία και χρειάζεται και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Πολλά κράτη-μέλη σήμερα προσπαθούν να αποδυναμώσουν, να στρεβλώσουν τη νομική βάση για το Σέγγεν και να αφαιρέσουν το δικαίωμα συναπόφασης του Κοινοβουλίου. Τι σκοπεύει να, κάνει η Πολωνική Προεδρία έναντι αυτής της απόπειρας. Είπε η Προεδρία ότι θα ήθελε η Ρουμανία και η Βουλγαρία να μπουν στο Σέγγεν Γνωμοδότησε ήδη σχετικά το Κοινοβούλιο. Τι σκέφτεται να κάνει η Προεδρία για να καταλήξει σε συμφωνία στο Συμβούλιο, κύριε Ρομέρο. Πρώτη ερώτηση. Εξωτερικά σύνορα και έλεγχη στα νότια σύνορα. Έρχομαι από την Ισπανία που μοιάζει πολύ με την Πολωνία που έχει και αυτή εξωτερικό σύνορο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ. Τι θα κάνετε για να καταργήσετε τις θεωρήσεις για ανθρώπους οι οποίοι, για τους οποίους είναι πραγματικά ντροπή και υποτιμητικό όλη αυτή η διαδικασία, καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμονες, ε, δικηγόροι, τέλος πάντων που θέλουν να κινηθούν, πώς θα, τους, ε, πώς θα το λύσετε αυτό. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση εσείς ε, θεωρείτε ότι μπορείτε να σμπρώξετε τη συμφωνία μέσα στο Συμβούλιο και θεωρείτε ότι στο επόμενο Συμβούλιο θα καταλήξετε σε μια συμφωνία για το ποινικό μέσο, δηλαδή η οδηγία που υπάρχει για το ποινικό ε, να αρχίσει να ισχύει είναι μια κατεπίγουσα οδηγία τη ζητάνε οι γυναίκες ανυπόμονα για το άσυλο. Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να διακρίνετε ποιον μηχανισμό θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε διάκριση μεταξύ της μετανάστευσης και του ασύλου ή θα πρέπει το Συμβούλιο και η Πολωνική Προεδρία να δώσουν μια Ό,τι, Δεν μπορούμε εμείς να συγκρίνουμε τους οικονομικούς μετανάστες με ανθρώπους που έρχονται από τραγωδίες. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς ε, που ήρθαν να μας παρουσιάσουν τις προτεραιότητες του σήμερα. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσεως και κατά την άποψή μου τέτοιου είδους περίοδοι ε, ε, είναι η περίοδοι κατά τις οποίες δείχνει κανείς αλληλεγγύη και δοκιμάζεται η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των ανθρώπων. Εγώ είμαι η συγγήτρια για την ε, αναδιατύπωση του Δουβλίνου 2 και όπως γνωρίζετε έχει κολλήσει εντελώς στο Συμβούλιο. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχετε σκοπό να κάνετε προκειμένου να ε, ε, ξεμπλοκάρει όλη η διαδικασία, να μπορούμε να προοδεύσουμε με το Δουβλίνο 2, με τον κανονισμό Δουβλίνο 2. Άλλωστε έχουμε και μια προθεσμία το 2012 και το χρωστάμε στους ε, πολίτες μας να τους προσφέρουμε αυτό που τους υποσχεθήκαμε το 1999 στο Τάμπερε και στη Στοκόλμη το 2009. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και ελπίζω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει ένα παράθυρο ευκαιρία η Πολωνική Προεδρία. Και καλή σας τύχη. Ευχαριστώ. Κύριε Ταβάρες, λέει ο Πρόεδρος. Δεν είναι εδώ πια. Ήταν στον κατάλογο παρόλα αυτά των ομιλητών. Τέλος πάντων. Κύριε Γιακολίνο. Θα είμαι πολύ πολύ γρήγορος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Υπουργούς. Σήμερα Έληξε και η προθεσμία για τις τροπολογίες σε δύο εκθέσεις εσωτερική απόσπαση εργαζομένων με, μεγάλη ειδικότητα από τρίτες χώρες και επίσης οι τροπολογίες για τους εποχιακούς. Ε, ρωτώ τον Υπουργό Εσωτερικών. Τι σκοπεύετε να κάνετε Προηγουμένως είπατε ότι θα έχουμε θετικές δράσεις υπέρ της Λαμπεντούζα, της Μάλτας, της Ελλάδας κλπ. Έναντι των βο... χωρών της Βορειοαφρικής. Ποιες θα είναι αυτές οι θετικές δράσεις? Κυρία Χέντ. Ο Υπουργός μίλησε για την προστασία των θυμάτων ε, των πιο δυνάμων θυμάτων ε, των εγκληματιών και σκέφτομαι εδώ τα παιδιά τα οποία είναι ιδιαίτε, παίζουν σημαντικότατο ρόλο κυρίως από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Για τα παιδιά, πρώτη ερώτηση. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στη βία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερον, παρότι τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει όλες τις συμβάσεις για την παιδική ηλικία, μόνο τα μισά από αυτά έχουν νομοθετήσει σχετικά. Θα συζητηθεί κάτι στο Συμβούλιο Υπουργών. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για τα δικαιώματα των παιδιών. Η κυρία Λάτφορντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να συμφωνήσω με άλλου συναδέλφου που έθεσαν το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Συλλήψεω. Ε, έχει λάβει πάρα πολλά τέτοια εντάλματα συλλήψεω στο Ηνωμένο Βασίλειο από πλευρά Πολωνία, αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτό. Ε, τονίσατε ιδιαίτερα το θέμα των ευρωπαϊκών αξιών και τη διατήρησή του. Ε, τι θα κάνετε λοιπόν ε, για το γεγονός ότι ε, θα μπορούσε το κάθε κράτος μέλος να αξιολογεί κάπως τις επιδόσεις του άλλου κράτος μέλος ε, για την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τη στιγμή που είμαστε όλοι μια Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα έπρεπε να παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν η πολωνική κυβέρνηση θα ενθαρρύνει τον Πολωνό εισαγγελέα να ολοκληρώσει την τετραετή ε, κράτηση και τα ε, βασανιστήρια που γίνονται σε ορισμένες φυλακές. Τέλος πάντων καταγγελίες που υπάρχουν σχετικά με αυτό το θέμα. Thank you for ε, this Η κυρία Μπάουερ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, σας... Ε, ρωτήσω σε σχέση με την αισιοδοξία για το μέλλον της ε, κοινή ε, πολιτικής ασύλου και επειδή η φιλοδοξία σας, η και η αισιοδοξία σας είναι πάρα πολύ εντυπωσιακέ, τι συμβιβασμό, τι λύση περιμένετε σε σχέση με το θέμα αυτό. Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ένα νομοθέτημα για την οικογενειακή βία κατά των ε, γυναικών. Αυτό έγινε σε προηγούμενες προεδρίες. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Πολωνική Προεδρία έχει σκοπό να το συνεχίσει. Η κυρία Μπλινκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς για την παρουσίασή τους και θα ήθελα να ευχηθώ για κάθε επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία. Έχω δύο ερωτήσει. Το πρώτο ερώτημα αφορά το πρόγραμμα απελευθέρωσης θεωρήσεων. Η Πολωνία έχει δεσμευθεί να ε, ε, παρέχει πλέον καλύτερες συνθήκες ε, για τις ανατολικές χώρες και αναφέρομαι κυρίως στην κατάσταση για τη, με τη Λευκορωσία. Ζητήθηκε από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστούν πιο εντατικά σε σχέση με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με τη χώρα αυτή ε, θα αναζητήσει μέτρα τέτοιου είδους η Πολωνία για τη Λευκορωσία, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένα ακόμη ερώτημα προς τον Υπουργό Μίλλερ πώς έχετε σκοπό να εξασφαλίσετε την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ε, σύστημα Σέγγεν. Και μία ακόμη ερώτηση προς τον κύριο Κφιατκόφσκι για τα μέτρα που αφορούν την οδηγία κατά των διακρίσεων, των μέτρων κατά των διακρίσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία, αλλά έχει κολλήσει και δεν υπάρχει συμβιβασμός. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κυρία Μπαντία. Ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ που ήρθατε να παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε προηγουμένως για την καταπολέμηση της τοξικομανίας. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε πραγματικά. Εντάξει για τις συνθετικές ουσίες, αλλά τι διάσταση θα δώσετε ακριβώς. Κύριος Παπανικολά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ κάθε επιτυχία στην Πολωνική Προεδρία. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το Δουβλίνο και το Eurodac και τους σχετικούς κανονισμούς. Οι ε, διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει εδώ και καιρό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έγιναν έτσι κάποιες, ε, υπήρξαν κάποια γεγονότα, είχαμε κάποιες ε, αποφάσεις για τον ε, κανονισμό Διβλίνου 2, είχαμε κάποιες μεμονωμένες αποφάσεις των κρατών μελών για διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτήν που προκύπτει από το Δουβλίνο 2. Η Πολωνική Προεδρία λοιπόν πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών θα έχουμε κάποια πρόοδο και ίσως ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει τώρα θα μπορέσει να άρει αυτό το αδιέξοδο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργή για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και για την πολιτική σας βούληση, για το πολιτικό σας μήνυμα το οποίο το στέλνετε πραγματικά σε μια πυρετόδη στιγμή της Ευρώπης εγώ θα στείλω ορισμένε γραπτές ερωτήσει στον κύριο Πινιατόφσκι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ποινικά. Θέλω όμως να ρωτήσω στον Υπουργό Εσωτερικών υπογραμμίζοντας αυτό που είπε και ο συνάδελφος Διέσδε Μέρα. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τον ανθρωπιστή συνάδελφο Γκέρεμεκ, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε νωρίς. Τι θα έλεγε πραγματικά για όλα αυτά. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να είστε ήσυχοι, κάντε ησυχία συνάδελφοι λέει ο Πρόεδρος. Οι συνάδελφοι έρχονται για την ε, ψηφοφορία, αλλά έχουμε ακόμα την ε, ακρόαση. Έχουμε προσκεκλημένους δύο υπουργού. Ε, σας ζητώ να κάνετε ησυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν. Παρακαλώ, συνεχίστε. Τι θα έλεγε λοιπόν ο κύριος Μέκα άμα έβλεπε ότι όλοι χαρήκαμε πραγματικά για την δημοκρατική πνοή στην Νότια Μεσόγειο και αν έβλεπε σήμερα την υποκρισία μας σήμερα αν έβλεπε δηλαδή πώς εμείς ε, ξαναπηγαίνουμε στη χώρα τους ε, ε, αυτούς που η μοίρα τους είναι τόσο τραγική. Τι θα κάνουμε λοιπόν για αυτές τις χιλιάδες πρόσφυγες. Κυρία Μακοβέη ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καλή τύχη στην Προεδρία σας. Τον Ιούνιο η Κομισιόν υιοθέτησε μία ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το κόστος της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μία, ένας ε, μηχανισμός υποβολής ε, εκθέσεων έχει μέσω αυτής της ε, απόφασης δημιουργηθεί και τώρα τον χτενίζουμε, χτενίζουμε τις λεπτομέρειες. Σας ζητώ λοιπόν να συμβάλλετε ώστε να προωθήσουμε αυτόν τον μηχανισμό και τον σχετικό στόχο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ελπίζω να έχουμε ένα ψήφισμα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο προς αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο, και τους δύο υπουργούς για, την, για το χρόνο που μας έχουν αφιερώσει σήμερα. Παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να ακούσουμε τις απαντήσεις των δύο Υπουργών. Ο κύριος Μίλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση είναι ε, κρίσιμη. Πρόκειται για μια ε, ε, πολύ σημαντική κρίση. Πώς θα βοηθήσουμε τη Μάλτα και την Ιταλία να τους βοηθήσουμε καταρχήν αυτούς που έρχονται στη Μάλτα και στην Ιταλία να μην έρχονται. Να τους βοηθήσουμε δηλαδή στις χώρες τους. Να προστατεύσουμε τα, τα ευρωπαϊκά σύνορα. Όσον αφορά στη συνεργασία με τις τρίτες χώρες στα πλαίσια του Σέγγεν. ποιο είναι το πρόβλημα για την Ευρώπη. Εάν κάποιος ε, παρουσιάσει ένα αίτημα, μια αίτηση ασύλου, αυτός που ζητάει το άσυλο μένει, παραμένει στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις τρίτες χώρες πρέπει όμως να έχουμε την συμφωνία επανεισδοχής. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου στις δικές μας χώρες να μπορούν να επιστρέφουν στις χώρες τους μετά. Για την Ρουμανία. Σας ευχαριστώ για την... και την Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ για την ενιαία θέση την οποία έχετε αναλάβει. Γνωρίζετε ότι η τελική λύση άπετη να εγκρίνουμε ομόφωνα το μέτρο αυτό. Γι' αυτό και παλεύουμε να περάσουμε αυτό το μέτρο. Ελπίζω σε μερικούς μήνες να μην μιλάμε μόνο με ευχολογίες, αλλά να μπορούμε να μιλάμε με συγκεκριμένα και χειροπιαστά πράγματα. για τους εποχιακούς. Εγώ δεν νομίζω ότι ως κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προστατευτούμε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλές μεγάλες ειδικότητες, είναι ιδιαίτερα ειδικευμένοι, δουλεύουν στις, σε, σε, σε επιχειρήσεις, σε σημαντικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ της Ευρώπης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε όλοι αυτοί οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να δουλεύουν στην Ευρώπη. Κυρίως σε αυτή τη φάση όπου θέλουμε οικονομική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο σε αυτή τη φάση. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις λύσεις. Για τους εποχιακούς εργαζόμενους γνωρίζουμε ότι χωρίς αυτούς τους εποχιακούς εργαζόμενους για ορισμένους κλάδους της οικονομίας θα έχουμε τεράστιες απώλειες. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε ανοιχτοί σε αυτού του τύπου της λύσης, γιατί κατά βάθος είναι καλό πράγμα. Αυτού του είδους η μετανάστευση, νόμιμη μετανάστευση, αυτό το οποίο κάνει είναι να ενισχύει την οικονομία και μειώνει το ρίσκο για την παράνομη μετανάστευση. Τώρα για την αισιοδοξία. Βεβαίω και είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι υπό την έννοια ότι θέλουμε να διευρύνουμε τις εργασίες για το πακέτο του ασύλου και αυτή την αισιοδοξία την έχουμε ακόμη περισσότερο όταν ξέρουμε ότι θα συνεργαστούμε με σας για την απολευθέρωση των ε, θεωρήσεων με τη Λευκορωσία. Μα είναι γειτόνι μας. Ε, δεν μπορούμε εμείς όμως να μεταχειριζόμαστε, ε, εμείς πρέπει μάλλον να μεταχειριστούμε με άλλον τρόπο τον κύριο Λουκασέγκο και αλλιώς τους, τους Λευκορώσους. Τώρα πώς θα το κάνουμε δεν ξέρω. Για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Γιατί μιλάμε. Για το πώς μπορούμε να μοιραστούμε το know-how. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να καταρτήσουμε τους υπαλλήλου που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών στις χώρες τους. Ξέρετε, οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά και η συνεργασία μας δεν θα πρέπει να γνωρίζει σύνορα, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Για την Eurodac και το Δουβλίνο, αν θα έχουν προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε. συζητάμε πια τόσο πολύ που θα πρέπει να δώσουμε λύσεις, κυρίως αυτή την εποχή κρίσης. Το είπαν αυτό όλοι. Σε περιόδους κρίσης πρέπει να είμαστε πιο αλληλέγγυοι. Και αν δεν το πετύχουμε, τότε δυστυχώς αποτύχαμε. Αυτά, πρόεδρε. Φανταστείτε τι θα γίνει όμω, ήδη από, τον πρώτο από την πρώτη μέρα έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, όταν θα ξανάρθω να δείτε τι θα κάνω. Λέει ο Ζητώ συγγνώμη. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι λίγο πιεσμένα πάντα. Ο Υπουργό Βιατκόφσκι έχει το λόγο. Ησυχία συνάδελφοι, ησυχία στην αίθουσα. Panie ναι, και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Όσον αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση για τα ποινικά. Μα ήδη έχουμε έναν οδικό χάρτη που εγκρίθηκε πίσω ειδική Προεδρίας για να αναπτύξουμε τα διαδικαστικά δικαιώματα ε, τις ε, διαδικαστικές φάσεις. Εδώ και 20 χρόνια παλεύουμε για το ποινικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δύο σχέδια. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των θυμάτων. Φυσικά, ε, για την οικονομική πραγματικότητα. Πρέπει να, να αξιολογήσουμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Για την κυρία Ρομέρο και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Εγώ ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε πριν η Κομισιόν παρουσιάσει αυτό το σχέδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ένταλμα σύλληψη, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Πολλοί μιλάνε για τη βία, την οικογενειακή βία και η Ισπανία έχει συνυπογράψει ε, ένα σχέδιο ε, το οποίο παρουσίασε για την καταπολέμηση της οικογενειακής βίας ε, υπό την Προεδρία της για τα παιδιά Πέρυσι στην Πολωνία εγκρίναμε ένα νόμο που απαγορεύει τη φυσική τιμωρία κατά των παιδιών. Είναι κάτι το οποίο με καίει πραγματικά και θα το συζητήσουμε και με άλλους υπουργούς δικαιοσύνης σε αυτή την Προεδρία. Για την για την για τις ανακρίσεις και τις έρευνες. Στην Πολωνία είχαμε τις σχετικές έρευνες για τις παράνομες κρατήσεις και ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας επίσης μου το επισήμανε. Η απόφαση η απόφαση για το θέμα της προφυλάκησης είχε ληφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση όταν είχαμε συζητήσει και το ρόλο του εισαγγελέα, του Γενικού Εισαγγελέα. Και ε, αυτός ο εισαγγελέα πλέον με τη μεταρρύθμιση είναι εντελώς ανεξάρτητος. Σε αυτό το πλαίσιο και η δική μου κυβέρνηση περιμένει την απόφαση για την ανεξάρτητη εισαγγελία όπως θα προκύψει από αυτήν την έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις τους, για την κατανόηση, για τις εξηγήσεις που μας έδωσαν, για την κατανόηση που έδειξαν στο πώς τρέχουν οι διαδικασίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Πραγματικά θα συνεχίσουμε την συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας. Οπότε θα σας ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ και τους δυο. cloud Please. Please. We're about to get started. Να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Take your seats. Καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι. Καθίστε, συνάδελφοι. Καθίστε. It's been some minutes of understandable delay as Εντάξει, έχουμε την ε, ακαδημαϊκή καθυστέρηση γιατί είχαμε εδώ τους ε, δύο υπουργού. Αλλά τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Δεν έχετε την κάρτα σας? Α, μπορείτε να τη βρείτε με κάποιο τρόπο. Ναι, Πρόεδρε, εγώ αντικαθιστώ τον ε, συνάδελφο. Ζήτησα για τη δική μου κάρτα την ηλεκτρονική, αλλά ακόμα δεν, δεν έχει έρθει. Ωραία. Οπότε θα προσθέτουμε κάθε φορά και έναν, μία ψήφο για τους σοσιαλιστές στον ηλεκτρονικό έλεγχο. Ελπίζω να μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέχρι να πάρετε την κάρτα σας. Υπάρχει κάποιος που να μην έχει την κάρτα του, η κυρία Γκρίσπεκ. Η κυρία Γκρίσπεκ από το Άλντε. Άλλος κανείς που να μην έχει την κάρτα του, ο κύριος Άλβαρο, την έχετε. Α, Mastercard είναι αυτή που έχετε. Α, όχι, Visa παίρνουμε μόνο. Μόνο Visa παίρνουμε. Η Mastercard δεν περνάει. No. Yes, yes, yes. Then, let's get started. Λοιπόν, ξεκινάμε για να μην καθυστερούμε πολύ. Πρώτη ψηφοφορία. Σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και παιδική πορνογραφία. Ψηφοφορία για την έκθεση της συναδέλφου Ρομπέρτα Αντζελίλη. Προτείνω να ακούσουμε σύντομα την εισηγήτρια να μας μιλήσει λίγο για την ε, ψηφοφορία, ίσως να μας ε, βοηθήσει αυτό να περιμένουμε να έρθουν και οι κάρτες που είναι στο δρόμο προς το παρόν. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ στο Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι ένα πολύ καλό κείμενο, μια πολύ καλή συμβαστική λύση που επετεύχθη μετά από εργόδη προσπάθεια, εννέα τριμερείς, διαλο... διαλόγους και θέλω να ευχαριστήσω ε, τους εκπροσώπους της Κομισιόν, του Συμβουλίου και τους Κιώδης ιδιαίτερα που δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να βελτιωθεί το κείμενο. Εκ μέρου λοιπόν των ομάδων θα ήθελα να ε, κάνω μια προφορική τροπολογία για τους, ε, κανόνες, για τους ε, πίνακες αντιστοιχίας. Αυτό το θέμα είναι προτεραιότητα για όλο το Κοινοβούλιο και έχει επιβεβαιωθεί δύο φορές μάλιστα από την διάσκεψη των Προέδρων. Προφανώς αυτό θα επισύρει κάποια προβλήματα, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να βρεθεί λύση εάν ε, το Συμβούλιο και η Προεδρία θέλει να βρει μια λύση. Το θέμα είναι να υπάρχει η βούληση. Χωρίς τους πίνακες αντιστοιχίας δεν θα γίνει αποδεκτή ε, η έκθεση από, τους, ε, από την διάσκεψη των Πρόεδρων για την Ολομέλεια. Οπότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την ισχυρή πολιτική επιλογή που έχει κάνει το Κοινοβούλιο για μας είναι προτεραιότητα να ψηφίσουμε για αυτή την οδηγία αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα, ένα οδηγό σύγκρισης για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αυτή την οδηγία και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που έχει υποβάλει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Καταλάβαμε, κυρία Αντζελίλη. Η συγκήτρια λοιπόν προτείνει να ψηφίσουμε unblock σε σύνολο το, την, την, ε, το κείμενο της ε, τροπολογίας 343 μαζί με την προφορική τροπολογία. Συμβαστικό κείμενο λοιπόν. 343. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ναι, ηλεκτρονικά, συγγνώμη. Άρχιδη ψηφοφορία. Now the Πέρας ψηφοφορίας. 50 ψηφίσαντες, 47 υπέρ, 3 αποχές. Βάζουμε μία συν για τους ε, σοσιαλιστές και δύο για τους ε, φιλελεύθερους. Οπότε, θα, οπότε είναι 49 υπέρ και 3 αποχές. Πολύ ωραία. Οπότε εγκρίνεται. 50, 50 υπέρ. Συγχαρητήρια κυρία Αντζελίλη. Now, now we, now we voting. Τώρα ψηφίζουμε Το σημείο 6. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας. Εισηγητής Ρούι Ταβάρες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Και πάλι 50 ένας ψηφίζαντες, 46 υπέρ, 1 κατά 4 αποχές, 2 υπέρ, 3 υπέρ. Όχι, όχι. Ε, εντάξει, ε, το, η σοσιαλιστική κάρτα βρέθηκε. Οπότε 2 για τους φιλελεύθερους, άρα 48 υπέρ, ένας κατά και τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Ταβάρες. Και στην Ισλανδία και στην Ορβηγία. We proceed. Thank Now, Τώρα. Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής εργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Frontex. Σάιμον Μποσούτιλ, ο εισηγητής. προτείνει και αυτός ε, ε, ψήφο unblock στο σύνολο για, την, ε, το κείμενο της, τροπολογία της τροπολογίας 255. Κύριε Μπουσούτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, προετοίμασα έναν λόγο μισής ώρας για να σας εξηγήσω. Αποκλείεται να πάρετε το λόγο για μισή ώρα, κύριε Μπουσούτη, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, όχι, απλώ ε, για να ευχαριστήσω όλου όσου συμμετείχαν στου τριμερεί διαλόγου και στη δουλειά που τελικά μα βοήθησε να καταλήξουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ήταν πολύ επιτυχέ το αποτέλεσμα και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του συναδέλφου από την Κομισιόν και το Συμβούλιο που ε, συνεργάστηκαν στον φάκελο αυτό, κυρίως όμως τους σκιώδεις συγητές που συνεργάστηκαν μαζί μου, που πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ να βελτιώσω το φάκελο αυτό. Ε, τέλος, να ευχαριστήσω τους συμβούλους μου, τους βοηθούς μου και την Helen Callors που είναι δίπλα σας για την ε, πραγματικά ανεκτήμητη βοήθειά της για το έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Και εμείς βεβαίω είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσους βοήθησαν. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία του συμβαστικού κειμένου όπως εξηγείται από τον κύριο Μπουσούτιλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ε, υπέρ, 53 ψηφίσαντες, 5 κατά και 7 αποχές. Οπότε μόνο ένα είναι από τους ε, φιλελεύθερους, άρα 42 υπέρ, 5 κατά και 7 αποχές. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται η έκθεση και συγχαρητήρια στον κύριο Μπουσούτιλ. 19 σελίδες τροπολογιών γλιτώσαμε, καταπληκτικά νέα. Και γι' αυτό κυρίως σας συγχαίρουμε. Ωραία, περνάμε τώρα στο σημείο 8 που αφορά την αντιδρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. Έχουμε εδώ τη συνάδελφό μας, Σοφία Ινετφέλτ, που είναι η συγγήτρια. Θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Απλώ θα ήθελα να πω ότι παρά το γεγονό ότι δεν συμφωνούμε σε όλα τα σημεία, θα ήθελα να αναγνωρίσω την προσπάθεια που έκαναν όλοι και ειδικότερα του Συμβούλους Πολιτικών και, τους, για ε, ε, βοηθό μου, το βοηθό μου κυρίως που περισσότερο από τον καθένα ε, του, αξίζει, του αξίζουν διακοπές. Μάλιστα. Αρχίζουμε λοιπόν τις συμβιβαστικέ τροπολογίες που μας κάνουν τη ζωή ευκολότερη και την ψηφοφορία ευκολότερη. Λοιπόν, συμβιβαστική 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τώρα. Καταπίπτουν πολλές τροπολογίες τότε και φτάνουμε. Στην ε, Γιούρι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αφέτ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την αφέτ 1. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 προς 30. Οπότε, περνάμε στην τροπολογία 83. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Φαινόταν σαν συμβιβασμό, αλλά εντάξει, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Άρχε ψηφοφορία. Πέρας. 29 προς 21 εγκρίνεται. Άρα, κάποιες καταπίπτουν και φτάνουμε στην τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικό στην 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 προς 23 εγκρίνεται. Τζούρι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άφετ 2. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Να ελέγξουμε. Ήταν σαφέ το αποτέλεσμα, αλλά ας το ξαναψηφίσουμε. Δεύτερο τμήμα της ΑΦΕΤ 2 ηλεκτρονικός. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 προς 16. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 88 καταπίπτει. Και άλλες καταπίπτουν. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 3. Ναι, παρακαλώ, θέλετε κάτι να πείτε. Μισό λεπτό να βάλω τα ακουστικά μου, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, θα έπρεπε ίσως να ψηφίσουμε και την 89 δεν λέμε ότι καταπίπτει άμα περάσει ο συμβιβασμός. Πράγματι, πράγματι είναι γραμμένο από κάτω. Οπότε ας περάσουμε πάλι στο... στην Γιούρι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικός για την Γιούρι 3. Πέρας. 35 προς 18. Άρα εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια για να βλέπουμε. Εγκρίνεται λοιπόν. Εκατό. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 Α, θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 106 Ωραία ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν πέρα της ψηφοφορίας. 14 37, άρα απορρίπτεται. 109 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 5, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ δεύτερο τμήμα ε, συγγνώμη κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς, δεν ήταν σαφές. Ψηφίζουμε την 103 ηλεκτρονικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 προς 33, άρα απορρίπτεται. Ωραία. Περνάμε στην 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά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 Ξέχασα την 138. Την ξέχασα. Καλά τα λέω. Ψηφίζουμε την 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αφέτ 5 υπέρ Α, όχι, θέλετε να ελέγξουμε τη Γιούρι 5? Ωραία να την ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός, άρχεται η ψηφοφορία. Now Πέρας, 20 προς 32, απορρίπτεται. Αφέτ 5, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ε, νομίζω ότι απορρίπτεται. Και αυτή. 119, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146-147 είναι ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γιούρι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άφετ 6 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 7. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα πάμε στη Γιούρη... Α, όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Την 158 πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 8. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, είπε κάποιος. Το δεύτερο τμήμα του Γιούρι 8. Τη τροπολογίας Γιούρι 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, απορρίπτεται. 19 προς 31. Άφετ 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιούρι 9. Α, όχι, ξέχασα την 162, λέει ο πρόεδρος. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιούρι 9 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άφετε 9, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163, 164, 165 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 10. Α, όχι, θέλετε να ελέγξουμε τις τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Ελέγχουμε ηλεκτρονικός άρχεται ψηφοφορία. We're voting. I mean, you know what, you know what we're voting? Okay, now closed. Πέρας ψηφοφορίας. 36 προς 15 κρίνεται. Γιούρι 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άφετ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167, 168 και 169. Αυτές είναι ταυτόσιμες και τις ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρί, ε, συγγνώμη, απορρίπτονται. 170 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171, 172 και 173 είναι τα... Α, συγγνώμη, λέει Πρόεδρος. Οι 171 και 172 είναι ταυτόσιμες και τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. αποχές. Απορρίπτονται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμπεβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γιούρι 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμπιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν κάποιες. Συμβιβαστική 18 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 188 δεν καταπίπτει και το ψηφίζουμε. Το δεύτερο τμήμα μόνο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193. Η Τζούρι 13 έχει καταπέσει. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμπεβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 14 υπέρ. Γιούρι 14, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε τη 201 ηλεκτρονικώς. Πολύ ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 201. 201. 201. Πέραση ψηφοφορία. 17 προς 31. Απορρίπτεται. Για 202 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 203. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 204. Κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 205 και 206 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 208 γιατί 207 έχει καταπέσει. Α, όχι, δεν έχει καταπέσει. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 210 καταπίπτει. Α. Ε, τότε 2.13 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται 214. Α θέλετε να ελέγξουμε τη 213 πρώτα. Ωραία, να την ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23 προς 27 απορρίπτεται. 214. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Αφετ 3. Καταπίπτει. Α, καταπίπτει. Η 215 όμως είναι ακόμη ζωντανή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217. Όχι, γιατί 216 πρέπει να ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρος. Μισό λεπτό. 216 τότε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 217. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 218 και 219 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 20. Έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 220. Καταπίπτει. Καταπίπτει. Mm. Ναι, αλλά αυτό δεν αναφέρεται στον κατάλογό μου. Άρα, 222 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 να ψηφίσουμε τη 222 ε, ας την ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίθηκε 33, 33 ψήφους προς 17 223 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. 224. Ελέγχουμε τη 224. Άρχεται η ψηφοφορία. Now closed. Πέρας. 29 προς 20 εγκρίνεται. And now the citations are recited. Πάμε σε ιδεολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. 14. 14. 14. 14? No. No. 14? No, oh, it's just, I mean, I got it fallen here. Μα αφού λέει ότι καταπίπτει. Then, then amendment 14. Favor. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω απορρίπτεται. Ε, να ελέγξουμε. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Πολλές καταπίπτουν. Πολλές καταπίπτουν. Πάμε στην 29. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Χωριστή ψηφοφορία λοιπόν. Πρώτο τμήμα της 29. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα της 29. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20. Favor. 20. 30. 30. sorry, I'm sorry. Yes, you're right. I'm sorry, I'm sorry. I'm also, I'm also, I'm also misleading the point here. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Παρανόησα εγώ. 30. Χωριστά σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34, 44, 44, 44 υπέρ. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 όχι. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει. 55. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59. 59 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60, υπέρ, κατά, Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνω. 60. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Εγκρίνεται. 61. Ε, α, καταπίπτει. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ 68 α συγγνώμη συγγνώμη ξέχασα τον 68 υπέρ λοιπόν για τον 68 κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ όχι, 70. Ουφ. Μα λέει καταπίπτει. Α. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Τέσσερα σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Όχι. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Τώρα Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 27 προς 24. Εγκρίνεται. 28 προς 24 γιατί έχουμε την ε, επιπλέον του Άλντε. 28 προς 24. Έχετε, είχατε πρόβλημα με, το, με την κάρτα σας. Εντάξει. Άρα συν 2. Άρα 29 προς 24. Εγκρίνεται λοιπόν. Εξακολουθεί να εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ενέτφελτ. Wow. We still have, we still have, please. Λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να έχετε εξαντληθεί πραγματικά, πρέπει να είστε πολύ κουρασμένοι, αλλά έχουμε άλλη μία έκθεση να ψηφίσουμε. Έχουμε άλλη μία έκθεση να ψηφίσουμε. So, please, please, I humbly, I humbly, I humbly request you. Σας ζητώ ταπεινά να μείνετε στην αίθουσα, να κάνετε ησυχία. Διαδικαστικό, κύριο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μπορώ να προτείνω την επόμενη, στην επόμενη συνεδρίαση να ζητήσετε μεγαλύτερη ε, αίθουσα. Γιατί δεν είναι λίγο η ατμόσφαιρα αποπνιχτική εδώ μέσα. Δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που το νιώθει αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε και μεγαλύτερη αίθουσα. Μακάρι. να είχαμε και άλλο χρόνο και άλλο χώρο και φρέσκο αέρα να είχαμε. Ωραία θα ήτανε. Θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πάντως για την πρόταση. Λοιπόν, ελάχιστα πρότυπα για, για το καθεστώς ε, των υπηκών τρίτων χωρών και των απάτριδων ω προσφύγων ή ω προσώπων που χρήζουν διεθνού προστασία καθώς και όσον αφορά το περιεχόμενο της εν λόγω προστασίας αναδιατύπωση. Η συγγήτρια Jean Lambert. Θέλετε το λόγο κυρία Lambert. Σύντομα όμως, ε. Ναι, ναι, ακούω ήδη τα μουγκριτά των συναδέλφων. Να ευχαριστήσω τους Κιώδης και όλους όσους συνεργάστηκαν για το έκθεση αυτή, γιατί δεν ήταν εύκολη. είπατε ότι όλοι έχουμε λίγο εξαντληθεί, ε, έχουμε κουραστεί πολύ και κάποιε από τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο μα έδωσαν την ίδια ακριβώ εντύπωση τη εξάντληση. Τώρα λοιπόν έχουμε μια συμβαστική λύση εδώ. Ελπίζω σήμερα το απόγευμα να μπορέσουμε να την εγκρίνουμε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και άλλο το πακέτο για το άσυλο. Υπάρχει μια τροπολογία, όπως με την κυρία Αντζελίλη, για το θέμα των πινάκων αντιστοιχία. Ε, Ελπίζουμε να, ελπίζαμε να είχαμε βρει λύση μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό. Παρόλα αυτά, στην τροπολογία μας, ε, τα άρθρα που αφορούν τους πίνακες, θα δείτε ποια είναι τα άρθρα που αφορούν τους πίνακες αντιστοιχίες, γιατί η αναδιατύπωση δεν είναι στο σύνολο μόνο, σε σύνολο μάλλον της έκθεσης, παρόλο που οι πίνακες ε, αντιστοιχίες για τα υπάρχοντα άρθρα νομίζω ότι θα ήταν εξίσου χρήσιμοι. Απλώς σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν εύκολο να υπάρξει συμβιβαστική λύση για το κείμενο αυτό μετά τις συζητήσεις με τους Σκιώδης, με, τους, με τον Τριμερή Διάλογο, με την Ουγγρική Προεδρία, την Κομισιόν και για το θέμα του, των πινάκων ε, αντιστοιχίας όντως έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες. Όντω λοιπόν δεν ήταν εύκολη δουλειά. Σα ευχαριστούμε για την συμβαστική αυτή πρόταση που έχουμε τώρα στο τραπέζι και πάμε στην ψηφοφορία. χωρίς καμία καθυστέρηση. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβιβαστικό κείμενο, ενοποιημένο, ψηφίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας για το συμβαστικό κείμενο. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε άρα στην τελική ψηφοφορία. Πολύ καλά νέα. Πάμε λοιπόν. Ε, ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Do we have? 45 υπέρ, 3 κατά. Μπράβο κυρία Λάμπερτ, ευχαριστούμε για το συμβασμό. Συγχαρητήρια. Τέλος οι ψηφοφορίες λοιπόν. Πάμε στο επόμενο σημείο.